και η βάση της πολιτικής μας. Και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλετε για την πολιτική γειτονία. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε δύο προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί. Μία για την ανατολική διάσταση της πολιτικής γειτονία και μία πρόταση ψηφίσματος για την νότια διάσταση τη πολιτική γειτονία. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12 η ώρα το μεσημέρι. Επόμενο ζήτημα, θέμα στην ημερήσια διάταξη, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρήση σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Τον λόγο θα λάβει και πάλι για την εξονομάτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Επίτροπος Φίλε και πάλι παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πρέπει με τους πιο αυστηρούς τρόπους, με, τους πιο, τα πιο αυστηρά λόγια να μιλήσουμε εναντίον της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Είτε πρόκειται για απλό εκφοβισμό, είτε πρόκειται για δεχθεί εγκλήματα. Πρόκειται για εγκλήματα που γίνονται εναντίον των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες ε, στον κόσμο, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, που δεν έχουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο προκειμένου να προστατεύσουν από τη βία τις γυναίκες και τα κορίτσια. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να ενθαρρύνει την υποβολή εκθέσεων για τέτοιες ε, επιθέσεις και δεν υπάρχει απαραίτητη νομοθεσία προκειμένου να αποθαρρυνθούν οι υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτές και προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ε, γυναίκες οι οποίες υφίστανται την έλλειψη αυτής της νομοθεσίας καθώς επίσης και πάρα, πολλές, πάρα πολλά ήθη τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στην κουλτούρα της κάθε χώρας. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Αιγύπτου βλέπουμε ότι είναι η θέση του άντρα αυτή η οποία προωθείται περισσότερο, ενώ δεν παρέχονται ίσα δικαιώματα στις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τιμήσουμε το θάρρο το οποίο έδειξαν οι γυναίκες από την Ισία και την Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Το ίμιση του πληθυσμού δεν συμμετέχει στον θεσμικό ανασχηματισμό. Καταλαβαίνετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση καταδικάζουμε τις παραβιές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά σεξουαλικές επιθέσεις, όσον αφορά τον βιασμό των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να ενδυναμώσει το ρόλο των γυναικών στην πολιτική, μη στρατιωτική, οικονομική ζωή και θα καταπολεμήσει σε κάθε περίπτωση τις διακρίσεις και την ατιμορρησία. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ των φύλων και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών. Στην διακήρυξη της Βαρκελόνης του 1995, σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, γίνεται ρητή αναφορά στην δέσμευση αυτή για την περιοχή της ε, Μεσογείου. Η ισότητα των ε, φύλων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες τις οποίες αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων στη διακήρυξη Βαρκελόνης το 2005 και κατά αυτόν τον τρόπο γιόρτσαν κιόλα την δέκατη επέτειο της ευρωμεσογειακής σχέσης. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης των Υπουργών αποφασίστηκε να ενδυναμωθεί ο ρόλος των γυναικών. Αυτό έγινε συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2006 στην Κωνσταντινούπολη. Και κατά αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε μία καινοτόμος πρόοδο στον τομέα αυτό. Υπουργοί από το Μαρόκο, την, το Λίβανο, από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, την Συρία και την Εσία συμφώνησαν να έχουν μια ολιστική προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις ακόλουθες αλλοσυνδεόμενες προτεραιότητες. Πρώτον, τα πολιτικά αστικά δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να προωθηθούν, θα πρέπει να έχουν τα, την, τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή, καθώς επίσης και την ίδια πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Έκτοτε από τη διάσκεψη του 2006 και μετά έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών και έχουν ιεραρχηθεί συγκεκριμένε προτεραιότητε, καθώ επίση και ένα μηχανισμό παρακολούθηση και έχουν γίνει συγκεκριμένε δημοσιεύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εταίροι λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μεσόγειο επαναβεβαίωσαν τι δεσμεύσει αυτέ στην δεύτερη διάσκεψη που έγινε στο Μαρακέ τον, Νοέμβριο του 2009. Η κοινωνία των πολιτών πάλι συμμετείχε πλήρω πλήρως συζητήσει που έλαβαν χώρα Αυξήθηκε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερο η ορατότητα του, προβλήματο του προβλήματος αυτού. Ήταν αυτό μια σημαντική πρόκληση με την οποία συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στην διάσκεψη αυτή. Πέρα από το περιφερειακό αυτό πλαίσιο, στον διμερή διάλογο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε, καθώ επίση και οι υποεπιτροπέ τη που έχουν να κάνουν με ζητήματα που άπτονται των δύο φύλων, είναι σημαντικά μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτέ οι σημαντικότατε ανησυχίε. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθεί τη βία κατά των γυναικών με οποιαδήποτε μορφή και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε θερμά, κύριε Επίτροπε. Περνάμε στου αγορητέ εξ ονόματο των κοινοβουλευτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Edith Μπάουερ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Thank so, so ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα το σθένος και την δέσμευση, έντονη δέσμευση του Επιτρόπου για την καταγγελία κατά δίκη της βίας κατά των γυναικών ως όπλο στις πολεμικές σειράξεις ε, που χρησιμοποιείται συστηματικά σε τέτοιες ένοπλες ε, σειράξεις ε, για την ταπείνωση, εκφοβισμό, πολιτική τρομοκρατία, απόσπαση πληροφοριών, η βία κατά των γυναικών σε ένοπλες σειράξεις βασίζεται σε παραδοσιακές απόψεις ότι οι γυναίκες είναι ιδιοκτησία των ανδρών. Εφόσον είναι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες διαβιβάζουν πολιτιστικά και παραδοσιακά τις αξίες η χρήση βίας κατά των γυναικών στρέφεται ουσιαστικά κατά της ίδιας της κοινωνίας και οι κανονισμοί του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναγνωρίζουν την βία κατά των γυναικών, σεξουαλική βία ως βία κατά του πληθυσμού διάφορες μορφές βίας σε ένοπλες σειράξεις που χρησιμοποιείται ο βιασμός, η ε, υποχρεωτική μέσω βιασμού εγκυμοσύνη, η, όλα αυτά παραβιάζουν τις αρχές της συμβάσης της Γενέβης και υπερβολικά συχνά η σεξουαλική βία σε περίπτωση πολέμου δεν τιμωρείται, δεν ε, ε, προσάγονται στη δικαιοσύνη οι ένοχοι. Ως τμήμα ακριβώς των εχθροπραξιών μένουν ατιμόρυτοι όσοι ακολουθούν, όσοι υιοθετούν τέτοιες πράξεις ε, είναι, ήρθε η χρονική στιγμή να καταδικαστούν αυτές οι απάνθρωπες πρακτικές οπουδήποτε στον κόσμο και το μήνυμα μας σήμερα πρέπει να είναι ότι οι υπεύθυνοι ένοχοι αυτών των εγκλημάτων πολέμου δεν μπορεί να μένουν ατιμόρυτοι, πρέπει να προσάγουν στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ, ξεπεράσει τον χρόνο σας, παρόλα αυτά σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες στην Προοδευτική Συμμαχία, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Αντίθετα με τις ε, πληροφορίες που φτάνουν τώρα από την Λιβύη, όπου βλέπουμε μόνο άντρες στην γραμμή, πρώτη γραμμή του πολέμου οι εικόνες στην κύρια πλατεία της ε, Βενγάζης ε, και σε σχέση και με διαδηλώσει διαδηλώσεις ε, στην Τινησία, στον Μπαχρέιν, στη Συρία, στην Ιορδανία έδειχναν γυναίκες όλων των ηλικιών που κράβγαζαν υπέρ της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Γυναίκες, κυρίως νέες γυναίκες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εκδηλώσεις αυτές, στις επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική. Η μοίρα αυτών των γυναικών που χαρακτηρίζεται από πατριαρχικές παραδόσεις παραδόσεις και θρησκευτικές παραδόσεις δεν είναι μόνο ενδεικτική αλλά καθοριστική για την πορεία που θα ακολουθηθεί τους επόμενους μήνες από αυτές τις χώρες αναζητώντας ε, την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις γυναίκες που με τόσο θάρρος ξεκίνησαν αυτές τις ε, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες ε, στην Άνοιξη, την Αραβική Άνοιξη. Να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών και να δοθεί υποστήριξη στις γυναίκες εκείνες που θέλουν ενεργά να συμμετάσχουν δίνοντας κίνητρα σε αυτές τις γυναίκες να συμμετάσχουν σε όλα τα δημοκρατικά όργανα και τα θεσμικά όργανα ως υποψήφιες κομμάτων, ως βουλευτίνες κτλ. Είναι απαραίτητο επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιήσει κάθε τι, ό,τι περνάει από το χέρι της για να καταπολεμήσει εκφοβισμούς και πρακτικές σεξουαλικές κατά των γυναικών που τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους. Όπως έχουμε την υποχρεωτική ε, αυτή ε, το θέμα της ε, Παρθενίας και βλέπουμε και την περίπτωση της ε, Λομπάιντι στην Λιβύη που είναι εγκλήματα που πραγματικά πρέπει να καταδικαστούν και βασιζόμαστε στο ότι είπατε εκπρόσωπος εσείς επίτροπε θα ζητήσετε άμεσα ανεξάρτητη διακρύβωση και εξέταση αυτών των περιπτώσεων ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ. Σας ευχαριστώ λέγει Πρόεδρος και τώρα για τους ε, ελεύθερους, φιλελεύθερους δημοκράτες θα λάβει τον λόγο η κυρία Παρβάνοβα παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή γιατί θέλαμε πραγματικά να μιλήσουμε για την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είδαμε α, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη και στην Αίγυπτο, ιδίω όσον αφορά τι γυναίκε. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επισέλθω σε λεπτομέρειε για όλε αυτέ τι περιπτώσει. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο συμβολικέ ενισχυτικέ καταστάσει που θα πρέπει να καταδικάσουμε αμέσω. Η Μαν Αλομπεϊντή, μία Λίβια, η οποία κατέθεσε σε δημοσιογράφου ότι διάστηκε ομαδικά από στρατιώτε και κρατήθηκε από τους στρατιώτες του Καντάφη και πέρασε από ανακρισία για πάρα πολλές ώρες πρωτού Στην Αίγυπτο πολλές διαδηλώτριες καταγγέλνουν ότι υποβλήθηκαν σε τεστ παρθενίας και βιάστηκαν από το στρατό και ορισμένοι τώρα δικάζονται για τις πράξεις αυτές. Ε, καταδεικνύουν όλα αυτά τα γεγονότα ότι ο βιασμό χρησιμοποιείται ακόμα σαν ε, πολεμικό όπλο κατά τον, του άμαχου πληθυσμού. Είναι απαράδεκτο εμείς να μην μιλήσουμε κατά των απέσιων αυτών ιδεχθών εγκλημάτων κατά των γυναικών. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αντιταχθούν και να, να, να στραφούν κατά της σεξουαλικής βίας και οποιασδήποτε άλλης κακομεταχείριση και κακοποίησης των, των γυναικών και όχι μόνο στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα απαραίτητα μέσα έτσι ώστε μετά την μετάβαση στις κοινωνίες αυτές οι γυναίκες θα έχουν τα θα, έχουν, θα, φέρουν, θα χαίρουν ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χθε μιλήσαμε περισσότερο για το ζήτημα τη ε, καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Σε καμία περίπτωση στα πλαίσια των πολιτικών μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχουμε ε, χαμηλότερα ε, πρότυπα από αυτά τα οποία έχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, αλλά και σε διάφορες άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχουμε ειδικέ πολιτικές υπέρ των γυναικών. Σε ευχαριστώ για τους πράσινους. Η κυρία Νοχμουδίρε, παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και για τα τεστ παρθενίας όσον αφορά τους Αιγύπτιους για τις γυναίκες που είχαν διαδηλώσει και την πολλαπλή, τον πολλαπλό βιασμό μιας Λίβιας υπηκόου από στρατιώτες η δεχτή συμβάντα αποτέλεσμα αυτού, αυτής της πρότασης ψηφίσματος. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να αυξηθεί αυτή η σεξουαλική βία αφενός στις σειράξεις στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό τον προηγούμενο Νοέμβριο εκφραστήκαμε υπέρ του ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση των γυναικών σε σειράξεις θα πρέπει επιτέλους να την πάρει στα σοβαρά. Εκπρόσωπος της ΥΠΑ της εκπροσώπου Άστον μίλησε τότε για τις πρόοδους που είχαν σημειωθεί υπάρχει μια, ένα βελτιωμένο πλαίσιο, διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών. Επιπλέον, πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει, έχουν εγκρίνει εθνικά προγράμματα δράσης με, την, με τις βέλτιστες πρακτικές best practices, πράγμα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα μέτρα και στον ε, ιατρικό τομέα, τομέα διέθεσε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ε, υιοθέτηση υλοποίηση αντίστοιχη πρόταση ψηφίσματο του ΟΗΕ. Και έτσι προβλέπονται και στρατηγικέ για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, καθώ επίση και η κατάρτιση προσωπικού σε περιπτώσει σειράξεων. Είναι ανάγκη τώρα όλα αυτά τα μέτρα ρητά και κατηγορηματικά στι ευρωπαϊκέ πρακτικέ για την γειτονία με τι χώρε του Νότου να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και να ληφθούν υπόψη. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου σίγουρα θα δοθεί από πλευρά μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ ευχαριστώ για την Ομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Φιγκερέδο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες έχουν ενεργά συμμετάσχει στι ε, επαναστάσει των πληθυσμών που ζητούν και διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε επίσης ότι αποτελούν μια πρακτική διαρκών ε, βιασμών και καταπίεση σεξουαλικής ε, εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα, εγκλημάτων πολέμου σύμφωνα με τη Σύμβαση τη Γενέβη και βλέπουμε ότι τα νέα τα οποία, οι ειδήσει οι οποίες ε, ε, που έχουμε από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, από την Λιβύη και από άλλες χώρες όπου υπάρχουν ένοπλες σειράξεις και πόλεμοι και γι' αυτό εμένουμε και επιμένουμε σε διπλωματικές αποτελεσματικές δράσεις που θα αντιστέκονται σε τέτοιου είδους ε, ομές βιοπραγίες σεξουαλικές, σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, οπουδήποτε αλλού. Υπογραμμίζουμε και χαιρετίζουμε τη σημασία να αναγνωριστεί ο ρόλο των γυναικών στι επαναστάσει και επιμένουμε στην ανάγκη να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή στι νέε δημοκρατικέ δομέ και νομικέ δομέ, οικονομικέ δομέ και πολιτικέ δομέ αυτών των κοινωνιών και να τερματιστούν οι αρνητικέ διακριτικέ μεταχειρήσει και αντιμετωπίσει των γυναικών που γινόντουσαν επί αιώνε εκεί. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Περνάμε στου επόμενου αγορητέ η κυρία Μπόσκορτ στη συνέχεια 1,5 λεπτό. Μπόσκορτ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η επανάσταση στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, οι επαναστάσει δίνουν ε, νέε δυνατότητε. Έχουμε την ευκαιρία να ανοικοδομηθεί δημοκρατία στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στου δρόμου ε, τη ε, Τίνιδα, ε, του Καΐρου και τη Μπενγάζη. Οι γυναίκε ήταν ένα σοβαρό στοιχείο, ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο όσον αφορά του ε, τα άτομα που διαμαρτυρόντουσαν. Έχουμε την περίπτωση βιασμού μιας νέας γυναίκας στη Λιβύη που ε, συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Δεν ήταν όμως οι μόνες ειδήσει ε, για την βία, για την βιασμού. Η βία χρησιμοποιείται ως όπλο κατά των γυναικών. Στο Κάιρο κακοποιήθηκαν γυναίκες για παράδειγμα από στρατιωτικούς. Στον πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο στην Λιβύη χρησιμοποιήθηκε πάλι η βία κατά των γυναικών, η βιασμή ως όπλο. Βλέπουμε σε μια κατάσταση ανομίας δεν υπάρχει υπάρχει καμία νομιμότητα, καμία, δεν, υπάρχει, κα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και οι γυναίκες είναι θυράματα της βίας. Ε, γι' αυτό πρέπει να εξεταστούν τέτοιες περιπτώσεις και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στα εγκλήματα αυτά. Πρέπει να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και ο ρόλος των γυναικών στην ανοικοδόμηση μιας ε, δημοκρατικής κοινωνίας δεν πρέπει να αμεληθεί. Θα πρέπει τα δικαιώματα των γυναικών να κατοχυρωθούν νομικά σε νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να βρουν τη θέση του οι γυναίκε στα κοινοβούλια, στι κυβερνήσει. Επίση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση είναι σημαντικά θέματα για τι γυναίκε. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τέτοιε πρακτικέ που αποκλείουν τι γυναίκε. Η ανεξαρτησία είναι σίγουρα η αιχμή του δόρατο για τι γυναίκε. και το επιχειρήν, η δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιχειρήσει και τα μικροδάνεια είναι πολύ σημαντική υπόθεση για τι γυναίκε. Στη συνέχεια παρακαλώ επόμενη αγώνα αγορήτρια Όιλαντ η ε, σεξουαλική επίθεση κατά των γυναικών αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κατά των ανδρών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή ανησυχούν ιδιαίτερα και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν από τις αρχές αυτών των περιοχών και από τις νέες δημοκρατικές δυνάμεις αλλά επίσης και από τα παλαιά καθεστώτα σχέση με αυτά θα ήθελα να υπενθυμίσω, να ζητήσω από την ύπατη εκπρόσωπο Άστον σε σχέση με την σεξουαλική βία σε αυτή την περιοχή αυτό να εξεταστεί με τους εκπροσώπους, αντιπροσώπους των ε, χωρών που εντάσσονται στην πολιτική γειτονία στις Ευρωπαϊκές Ένωσης ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι, οι υπεύθυνοι και να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των γυναικών και των ανδρών. Αυτή η μορφή βίας ε, είναι το χειρότερο όπλο που πρέπει να αποφεύγεται με οποιοδήποτε αντίτιμο και πρέπει να <clears throat> τιμωρούνται σκληρά οι ένοχοι. Αυστηρά η Ένοχη. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch Δύο αγορητέ, Σον Κέλλη και η κυρία Ζαμπόσκα μετά. Ο κύριο Κέλλη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Πριν από δύο μήνες μιλούσαμε για την βία εναντίον των γυναικών στην Ευρώπη και αναφέρθηκε τότε ότι γύρω στο 25% των γυναικών υφίστανται βία μέσα στην Ευρώπη. Τώρα μιλάμε για τη σεξουαλική βία εναντίον των γυναικών στις ε, συγκρούσεις στην ε, Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Είναι φρικτές ιστορίες που δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε πλέον. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε την κατάσταση αυτή είναι κάτι που αφορά ε, μια ολόκληρη Ήπειρο, την Αφρική. Συμφωνώ όμως με τον Επίτροπο ότι θα πρέπει να τονίσουμε το πρόβλημα αυτό και ιδιαίτερα να καταστήσουμε υπόλογους τους δράστες αυτών των εγκλημάτων με την ελπίδα ότι κάποτε θα αλλάξουν οι τροπίες και θα σταματήσει αυτή η αποτρόπαια κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαμπόσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Η σεξουαλική βία δεν είναι απλώς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για άντρες, είτε πρόκειται για γυναίκες. Ε, είναι μία βία η οποία τάσσεται κατά της αξιοπρέπειας ε, είτε των ανδρών είτε των γυναικών. Και αυτό σε οποιαδήποτε χώρα της ε, Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής. Στις εμβόλεμες διενέξεις δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την εμφάνιση των ε, ε, γεγονότων αυτών. Είδαμε ότι ε, έχουμε περιπτώσει βιασμού όχι μόνο κατά των γυναικών αλλά και των ανδρών. Θα πρέπει να αναλυφθεί απαραίτητη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξαφανιστούν τα φαινόμενα αυτά παντού παγκοσμίω. Θα πρέπει επίση να βρούμε ποια είναι τα απαραίτητα μέσα τα οποία θα μα επιτρέψουν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των γεγονότων αυτών και να καταφέρουμε να ελοποιήσουμε την πραγματοποίηση των αυτών των δικαιωμάτων. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Φίλε τώρα πάλι εξ ονόματο τη Επιτροπή. Παρακαλώ κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, τα ερωτήματα για συγκεκριμένες περιπτώσεις που θέσατε υπόψη μας απόψε είναι πραγματικά μια μελανή κοιλίδα ε, στα πλαίσια των πρόσφατων εξελίξεων των τελευταίων εβδομάδων στην Βόρεια Αφρική και στην ε, ε, Μέση Ανατολή. Σημείωσα όλα τα θέματα που θίξατε κατά τη συζήτηση αυτή και τις προτάσεις που διατυπώσατε. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορα μέσα και θα κάνει το ΠΑΝ για να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και ε, σε μια ε, πολιτική ζωή ελεύθερη από κάθε είδους ε, εκφοβισμό και βία. Επίσης θα ήθελα να σας ε, θέσω υπόψη κάποιες θετικές πρόσφατες εξελίξεις όπως ε, το, τη δημιουργία του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις χώρες συνεργασίας του κόλπου, στη γραμματεία της συνεργασίας αυτής. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοια βήματα. Επίσης, ε, θα πρέπει η υποστήριξη της διεθνής, της διεθνούς κοινότητας, των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Ε, θα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ε, και θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να συνεχιστεί με τους νέους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, πέντε προτάσεις ψηφίσματος κατατέθηκαν από πέντε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες. Τους πράσινους, της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών, το, της